κανόνων, μια ανοιχτή και δημοκρατική συζήτηση που κανένα δεν ήθελε να περιορίσει. Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα να την περιορίσω. Σα ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία τώρα. Παρακαλώ, αρχίζουν οι ψηφοφορίε. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη ψηφοφορία ε, για την έκθεση Μπέκε με θέμα την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του έργου ΙΤΕΡ. Ε, προφορική τροπολογία. Ο κύριος Λαμασούρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος Επιτροπής Προϋπολογισμών θα παρακαλούσα πριν ε, γίνει η ενιαία ψηφοφορία να θέσετε προς ψήφιση μια τροπολογία που εγκρίθηκε χτες το βράδυ ομόφωνα από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Είναι μια όψιμη ε, τροπολογία και για λόγους χρόνου δεν προλάβαμε να τη μεταφράσουμε σε όλες τις γλώσσες. Δεν μπορούσαμε όμως να πράξουμε διαφορετικά και πολιτικά είναι πάρα πολύ σημαντική η τροπολογία αυτή γιατί μετά τη συμφωνία που επετέφθη στον τριμερή διάλογο την περασμένη εβδομάδα για τη χρηματοδότηση του έργου ΙΤΕΡ το Συμβούλιο, και αυτό το μάθαμε χτες το απόγευμα, ενέκρινε ομόφωνα τη συμφωνία αυτή με μονομερή δήλωση που υπογράφουν όμως έξι κράτη-μέλη και δίδουν αντίθετη ερμηνεία ε, τα κράτη αυτά στη συμφωνία από την ερμηνεία που έδωσε την προσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό θεώρησε σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Προπολογισμών σήμερα το Κοινοβούλιο επίσημα ε, να ε, τοποθετηθεί. αλλιώς δεν θα είχαμε συμφωνήσει στο τριμερή διάλογο. Σύμφωνα με το άρθρο 161 εδάφιο 3 του κανονισμού μας μπορεί να τεθεί σε ψήφιση αυτή η τροπολογία έστω και όψιμη γιατί είναι έκτακτες οι σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών ζήτησε να ψηφίσουμε τώρα κάποιες ε, τροπολογίες ε, ερμηνείες που χθες εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα ήθελα πρώτα να σας ρωτήσω, είναι κανείς ε, ενάντια σε αυτή τη διαδικασία? Όχι, δεν υπάρχουν στάσεις για τη διαδικασία. Οπότε θα ψηφίσουμε αυτά που μας επισήμανε ο κύριος Λαμασούρ. Τη χθεσινή δηλαδή συμφωνία και τις τροπολογίες που υπερψήφισε χθες η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ποιος είναι υπέρ της χθεσινής συμφωνίας της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Παρακαλώ, διανατάσεις χειρός, κατά, αποχές, ωραία εγκρίθηκαν οι προτάσεις ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Επικυρώθηκαν και από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία της έκθεσης Μπέγκε. Με ονομαστική κλίση, μαζί με την τροπολογία που πριν από λίγο υπέβαλε ο κύριος Λαμασούρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και ευχαριστούμε τον κύριο για τον εισηγητή. Επόμενη έκθεση είναι η έκθεση για την Γεντζεγεύσκα, σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθμός 7 του 2011 για το δημοσιονομικό έτος 2011. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Γιαντζογεύσκα. Επόμενη έκθεση του κυρίου Μπέγκε για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Μπέγκε. Επόμενη έκθεση είναι η έκθεση της κυρίας Ματέρα για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση Ματέρα και ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Ψηφίσουμε την έκθεση ΣΥΠΕΛ για το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και η έκθεση ΣΥΠΕΛ και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Σέντερ, Αγιάλα Σέντερ, για τον διορισμό μελών του ελεκτικού συνεδρίου. Πρώτη ψηφοφορία αφορά το διορισμό του κυρίου Κάρελ Πίνξτεν. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ θα έχουμε μυστική ψηφοφορία. Μόνο ένα φως θα ανάψει, το γαλάζιο φως θα ανάψει στο μηχάνημά σας. Δεν θα φαίνεται δηλαδή αν ψηφίζετε υπέρ κατά ή αποχή. Η ψηφοφορία γίνεται κανονικά. Απλώς επειδή είναι μυστική ψηφοφορία θα ανάψει μόνο ένα γαλάζιο φως στο μηχάνημά σας. Ψηφίζουμε λοιπόν για το διορισμό του κυρίου Κάρελ Πίνξτεν στο ελεγκτικό συνέδριο. Άρχεται η συνεδρίαση. Άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ο διορισμός του κυρίου Πίνξτεν. Τον συγχαίρομαι. Ψηφίσουμε τώρα για το διορισμό του κυρίου Χένρικ Ότμπο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και ο διορισμός του κυρίου Ότμπο. Συγχαρητήρια. Ψηφίζουμε για το διορισμό του κυρίου Χουάν Φρανσίσκο Κορώνα Ραμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Διαπιστώνω ότι υπάρχει μια πρόταση του κυρίου Οντί. Ναι, κύριε Πρόεδρε. διεξάγονται διαβουλεύσεις για το διορισμό των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου. Θυμίζω ότι απαρτίζεται από 27 μέλη το άρθρο 186 ή 286 της συνθήκης ε, ορίζει ότι ε, είναι συμβουλευτική η ε, πρόταση του Κοινοβουλίου. Οι κυβερνήσεις προτείνουν ονόματα και το Κοινοβούλιο γνωμοδετεί. Έχουμε ένα σύνολο μελών, 8 από 8 χώρες, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Σουηδία. Μεταξύ των 8 αυτών κρατών, 4 έχουν αλλάξει κυβέρνηση. Ε, Βέλγιο, Ιταλία, Δανία και Ισπανία. Δύο με εκλογές, δύο χωρίς εκλογές. Ε, Βέλγιο και Ιταλία χωρίς εκλογές, με εκλογές Δανία, Ισπανία. Από τις τέσσερις αυτές χώρες, η μία στο βασίλειο της Ισπανίας είδε να αλλάζουν και οι πολιτικές δυνάμεις. Εγώ ήμουν στη Μασαλία στη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ. Τα υπόλοιπα τρία κράτη δεν έχουν ζητήσει τίποτα. Η Ισπανία και οι ισπανικές πολιτικές δυνάμεις μου ζήτησαν να παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναβληθεί, όπως προβλέπει το άρθρο 108 του εσωτερικού μας κανονισμού, να αναβληθεί η ψηφοφορία για να υπάρχει χρόνος ε, ο ε, Βασιλέα θα ορκίσει την κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα. Ε, το ζητεί λοιπόν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και υπάρχει δυνατότητα να αναβληθεί η ψηφοφορία. Sorry. Με βάση τον κανονισμό θα ήθελα να ζητήσω πρώτα ε, μία ε, ομιλία υπέρ του αιτήματο και μετά μία κατά. Ποιος θέλει να ε, μιλήσει υπέρ του αιτήματο του κύριο Ο κύριος Περόνι. Ευχαριστώ. Εν συντομία θα ήθελα να πω ότι στην Ευρώπη ε, μερικές φορές αγνοείται η βούληση του, του λαού. Είπαμε, στην Ελλάδα σχετικά πιέσει κατά του δημοψηφίσματος. Στην Ισπανία είχαμε πιέσει, στην Ιταλία ε, επίσης βέβαια. Ε, μετά τις εκλογές αλλάζουν ε, τα αποτελέσματα, γι' αυτό γίνονται και εκλογές είμαι υπέρ τη αναβολής γιατί η νέα ισπανική κυβέρνηση που, είναι, που βγήκε από τις ελεύθερες εκλογές θα επιβεβαιώσει ή θα προτείνει διαφορετική υποψηφιότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό της δημοκρατίας. Καλώ. Θα ήθελα τώρα κάποιο να μιλήσει κατά του αιτήματο, ο Αντιπρόεδρος ε, Σόβοντα. Πρόεδρε, Πέρα από το γεγονό ότι έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην εισηγήτρια κυρία Γιάλα Σέντερ, θα ήθελα να διαπιστώσω το εξή εξ ονόματο τη ομάδα μου. Η θέση αυτή είναι ανεξάρτητη. Είναι ένα πρόσωπο που είτε θεωρούμε σωστό είτε θεωρούμε λάθο. Δεν είναι εκπρόσωπο κάποια κυβέρνηση εντεταλμένο και θα πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα. Την επόμενη φορά Δεχομένω θα θελήσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να αλλάξει επίτροπο γιατί άλλαξε η κυβέρνηση. Εμεί στην Ευρώπη εκπροσωπούμε και όχι με μονομένε κυβερνήσει. Παρακαλώ να ληφθεί υπόψη αυτό. Και θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι εδώ διορίστηκε κάποιο, η Επιτροπή του Κοινοβουλίου το θεώρησε σωστό και δεδειγμένο το πρόσωπο. Η συγγήτρια κυρία Γιάλα Σέντερ ε, τα παρουσίασε όλα αυτά, οπότε κανονικά και σοβαρά θα πρέπει να ψηφίσουμε το πρόσωπο αυτό και όχι εκ των υστέρων για την κυβέρνηση στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε πρώτα το αίτημα του κυρίου Οντί που ζήτησε αναβολή της ψηφοφορίας για το διορισμό του κυρίου Κορώνα Ραμών. Πρώτα λοιπόν θα ψηφίσουμε το αίτημα του κυρίου Οντί. Ποιος είναι υπέρ του αιτήματος ε, του κυρίου Οντί. Θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε, επαναλαμβάνω, ε, ως προς το αίτημα του κυρίου Οντί. Ψήφισα όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το αίτημα Οντί. Οπότε ψηφίζουμε τώρα για το διορισμό του κυρίου Κορώνα Ραμών στο ελεκτικό συνέδριο. Μυστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Κανδιδατούρα Εγκρίνεται ο διορισμός του κυρίου Ραμών. Συγχαρητήρια. Διορισμός του κυρίου Βίλε Ήταλα για το ελεγκτικό συνέδριο. Μυστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ο διορισμός του κυρίου Ήταλα. Συγχαρητήρια. Επόμενος είναι ο διορισμός ε, του κυρίου Κέβιν Κάρντιφ. Άρχεται η μυστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και ο διορισμός του κυρίου Κάρντιφ. Επόμενος διορισμός του κυρίου Πιέτρ Ρούσο. Άρχεται η ψηφοφορία. Czy wszyscy głosowali? όλοι. Zamykam głosowanie. Εγκρίνεται ο διορισμός του κυρίου Ρούσο. Σε χαρητήρια. Διορισμός του κυρίου Βιτόρ Μανουέλ Ντασίλβα Καλντέιρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τι Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ο διορισμός του κ. Καλτέρα. Συγχαρητήρια. Και τελευταίος, τελευταία υποψηφιότητα του κυρίου Hans Gustav Βέσμπεργκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε και ο διορισμός του κυρίου Βέσπερκ και συγχαίρω την κυρία Σέντερα Γιάλα για την εκπόνηση όλων αυτών των εκθέσεων. Επόμενη έκθεση είναι ε, της κυρίας Χιμένες και της κυρίας Ρομέρο. Δεν υπευλήθηκαν αιτήματα ούτε απόρριψης ούτε τροπολογίας. Η κυρία Τέισεν ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να επανορθώσω κάτι που ακούστηκε λάθος. Ίσως δεν πίνω συχνά καφέ με τον συνάδελφό Ντι, αλλά η νέα κυβέρνηση του Βελγίου ήταν κατόπιν εκλογών. Χρειαστήκαμε πάνω από 500 μέρες για να σχηματίσουμε κυβέρνηση, αλλά ήταν η κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε. Ναι, ναι. Το γνωρίζουμε, αλλά καλά κάνατε και το υπογράμμισετε. Έχει νόημα. Γιατί η δημοκρατία χρειάζεται μερικές φορές χρόνο, αλλά τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Επανερχόμαστε λοιπόν. Δεύτερη ανάγνωση για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Έκθεση Χιμένες και Ρομέρο. Δεν ε, έχει υποβληθεί ούτε αίτημα απόρριψης της σύστασης ούτε τροπολογίες. Οπότε θεωρώ ότι γίνεται δεκτή η κοινή θέση του Συμβουλίου. Επόμενο θέμα, έκθεση Ματιού. Πάλι πρόκειται για σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση με θέμα τη διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας. Ούτε και εδώ έχουν υποβληθεί αιτήματα απόρριψης ή τροπολογίες. Οπότε θεωρώ ότι η κοινή θέση του Συμβουλίου εγκρίνεται. Και ευχαριστούμε την κυρία Ματιέ. Επόμενη έκθεση του κυρίου Ριβελίνη. Πάλι πρόκειται για σύσταση δεύτερης ανάγνωσης. Κάποιες διατάξεις ε, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο. Ούτε και εδώ είχαμε έτοιμα απόρριψης και καμία τροπολογία. Οπότε θεωρώ ότι η κοινή θέση του Συμβουλίου γίνεται δεκτή και ευχαριστούμε τον εισηγητή μας τον κύριο Ριβελίνη. Επόμενη ψηφοφορία, σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση με θέμα τους ετήσιους λογαριασμούς εταιριών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες. Πρόκειται για έκθεση του κυρίου Λένε. Εξετάζουμε τη θέση του Συμβουλίου. Έχουν κατατεθεί πέντε τροπολογίες από την Νομική Επιτροπή. Τις ψηφίζουμε από κοινό. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, εγκρίνονται μάλλον. Οπότε τροποποιείται το τρόπος η κοινή θέση. Σας ευχαριστώ και συγχαίρω τον εισηγητή μας τον κύριο Λένε. Επόμενη έκθεση είναι έκθεση του κυρίου Ντεκάστρο για ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση ορισμένων κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ή απειλούνται με σοβαρές δυσχέρειες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Εξετάζουμε το σχέδιο κανονισμού. Ψηφίζουμε το σύνολο των τροπολογιών, τις έξι δηλαδή τροπολογίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε τώρα την ούτως τροποποιηθήσα πρόταση Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Δεκάστρο. Και έχουμε τώρα την έκθεση Sturdy. Ε, σχέδιο ψηφίσματος. Παράγραφος 24. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η παράγραφος 24. Αιτιολογική σκέψη G. Κατά τμήματα. Τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη L. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη M. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη N. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη O. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίσουμε τώρα ολόκληρο το σχέδιο ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και ευχαριστούμε τον κύριο Στέρδη και σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. τους ε,